συνεχίσουμε αύριο. Περνούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξη κοινή συζήτηση για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Ε, the next... Το επόμενο θέμα είναι η κοινή συζήτηση για τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη. Έχουμε τις δηλώσεις ε, της, ε, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το Διεθνές ε, Συμβούλιο για τη Χρηματοδότηση και την Ανάπτυξη και την έκθεση της κυρίας Σλάιν για την φόρο αποφυγή και την φόρο διαφυγή ως προκλήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και ξεκινάμε τη συζήτηση με την εισηγητρία. Την κυρία Σλάιν. Έχετε το λόγο. Για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής ε, επίσης έχει τεθεί σε επίπεδο ε, Αντιμετώπιση και έχει καταστεί προτεραιότητα γιατί πολλές ε, κεφαλαϊκές ροές ε, μεταγκαταστούνται με ένα κλικ του ποντικού από ένα μέρο του κόσμου σε ένα άλλο. Αυτό είναι παγκόσμιο προκλήσει και θα πρέπει ω τέτοιε να τι αντιμετωπίσουμε γιατί θα πρέπει να ακολουθήσουμε αρχέ αρχές, μια απλή αρχή. Ο φόρο θα πρέπει να καταβάλλεται εκεί που γίνεται το κέρδο, εκεί που προσφέρει η υπηρεσία ή το προϊόν και θα πρέπει αυτό να έχει ένα, μια συνέπεια και για τις μελλοντικές γενιές. Η αλλαγή του κλίματος σε ό,τι αφορά θα το στήσω επίκεντρο της διάσκεψης της Αντισαμπέμπας και αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν μόνο αν υπάρχει σωστή χρηματοδότηση. Και με καλύτερη κινητοποίηση των εσωτερικών πόρων. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή και φορο, φοροαποφυγή. Υπολογίζεται ότι οι παράνομες οικονομικές ροές ε, στις αντισόμενες χώρες είναι ε, ένα δις ε, το χρόνο. Μιλάμε για πόρους που τους κλέβουμε από τους πολίτες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μην ξεχνάμε ότι Υπάρχει επίσης και φοβερός φορολογικός ανταγωνισμός που είναι επιζήμιος για τις χώρες αυτές. Με αυτή την έκθεση ζητάμε από την Κομισιόν ένα πραγματικό πρόγραμμα δράσης για να υποστηρίξουμε τις αντισώμενες χώρες. Σας παρακαλώ μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο ήρεμα. Ζητάμε από την Κομισιόν μια, ένα πραγματικό σχέδιο δράση για να υποστηρίξουμε τι αναπτυσσόμενε χώρε, για να, δημιουργήσουμε, να δημιουργήσουν πιο ε, δίκαια φορολογικά συστήματα. Να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτέ τι χώρε με τεχνική και οικονομική ε, στήριξη που δεν δίδεται επαρκώ. Ζητάμε ε, την μετατροπή ε, της, Επιτροπή του ΟΗΕ για τη φορολογία σε ένα πραγματικό οργανισμό ούτω ώστε να εξασφαλίζει ότι οι χώρες αυτές ε, συμμετέχουν επίση όρει στην μεταρρύθμιση για την παγκόσμια, στην παγκόσμια μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματο. Ε, όπως παραδείγματο χάρη το σύστημα BEPS που προωθεί ο ΩΣΑ. Θα πρέπει να λάβουμε πιο πολύ όμω ε, υπόψη τις ανάγκες των αντισωμένων χωρών. Με δύο εργαλεία υπόψη. Ζητάμε να υιοθετηθεί το πρότυπο του Country country reporting, δηλαδή ε, για όλες τις πολυεθνικές ε, ειδικές εκθέσεις αναχώρας και αυτές οι εκθέσεις να είναι δημόσιες για, και να αφορούν όλες τις χώρες. Θα μου έκανε εντύπωση αν αύριο κάποιο καταψήφιζε αυτό που υποστηρίξαμε ομόφωνα στην Κομισιόν. Επίση, όταν εφαρμόζεται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, θα πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδο για τι χώρε που δεν έχουν ακόμα αναπτύξει πλήρω το απαραίτητο δυναμικό για να δεχτούν και να μοιραστούν όλε τι πληροφορίε που του ζητάμε. Θέλουμε διαφάνεια για τις ε, διάφορες επιχειρήσεις, τα trust, δηλαδή τα καταπιστεύματα κτλ. Επίσης ε, θέλουμε ισοτιμία ανάμεσα στις ε, αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει ένα μοντέλο του ΟΗΕ για να λαμβάνουμε υπόψη με πιο δίκαιο τρόπο τα δεδομένα των όλων των χωρών. Πρέπει να υπάρχει ε, μια ισορροπία, ισορροπημένη πολιτική για την ανάπτυξη. Επίσης, θα πρέπει να, να, μέχρι το 2015 θα πρέπει να έχουμε μαυροπίνακα και κυρώσεις για τους φορολογικούς παραδείσους. Δεν θέλω να ψηφίσουμε διαφορετικά. νομίζω ότι όλοι είμαστε εδώ σύμφωνοι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με σοβαρότητα. Τελευταίο αλλά σημαντικό. Δίνουμε μεγάλη σημασία στα θέματα του φύλου. Ε, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή ε, πλήττει κυρίως τα πιο αδύναμα κομμάτια τη κοινωνία και προφανώ συχνά τι γυναίκε ω γυναίκες ως πιο αδύναμε. Ευχαριστώ το γραφείο μου, ευχαριστώ την γραμματεία και ελπίζω ότι αύριο θα περάσει αυτή η έκθεση με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία για να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου και να δείξουμε ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή του πυρό για την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγή. Για να δείξουμε την ε, φιλοδοξία μας και να αντιμετωπίσουμε το δράμα της φτώχεια και της ε, ανισότητας. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του Συμβουλίου έχουμε τον Υπουργό Σμίτ, ο οποίος έχει το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βουλευτές, Σχεδόν δύο χρόνια τώρα έχουν περάσει που εμπλεκόμαστε σε μια περίπλοκη διαδικασία διαπραγματεύσεων με στόχο μια παγκόσμια εταιρική σχέση για να ανταποκριθούμε στη πρόκληση της εκρίζωσης ε, της στόχιας ε, και της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι δύο άρρηκτα συνδεδεμένοι στόχοι. Για τις επόμενες χρονιές η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, διότι είναι ιστορικής σημασίας αυτή η εταιρική σχέση που πρέπει να βασίζεται στην αρχή της οικουμενικότητας, της κοινή ευθύνη και της αλληλέγγυας ευθύνη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ικανότητες ε, των εταίρων ε, και ε, να συνεργαστούν επίσης πολλοί άριθμοι εταίροι. Μέσα σε αυτή την εταιρική σχέση θα πρέπει να προωθήσουμε επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την μη διακριτική μεταχείριση, τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, την ορθή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Έτσι θα μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν ενεργά εξασφαλίζοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και το σεβασμό των περατών ορίων του πλανήτη μας, τα δικαιώματα των γυναικών, η χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών που είναι και αυτοσκοπή ε, συνιστούν όμως και απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση των προγραμμάτων μας και πρέπει να ενθαρρύνονται σε όλα τα επίπεδα. Σκέφτομαι συγκεκριμένα την ανατροφή των κοριτσιών που για στους στόχους της ανάπτυξης έχει ιδιαίτερη σημασία. Ε, μετά από τις πρώτες βάσεις της εταιρικής σχέσης χρειαζόμαστε ένα σφαιρικότερο όραμα που προσαρμόζεται στις παγκόσμιες αλλαγές. Η διάσκεψη στην Αντίσα που ξεκινά την επόμενη Δευτέρα δεν πρέπει να περιοριστεί σε έναν απολογισμό ε, της πρόοδου σε σχέση με το Μοντρέ και την πρόοδο που έχει ε, σημειώσει σημειωθεί αλλά θα πρέπει να οδηγηθεί στην ολοκλήρωση ε, και την ε, συσσόρευση όλων των μέσων ε, και οικονομικών και άλλων πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας για την εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να επιβεβαιώνουν αυτήν την βασική αρχή σε σχέση με τους δημοσίους πόρους που είναι η σταθερότερη και πιο εύκολα διαθέσιμη πηγή χρηματοδότηση και άρα βρίσκονται στην καρδιά της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών φέρουν την πρώτη στη ευθύνη για την κινητοποίηση και την χρηστή διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Μετά από αυτή τη διάσκεψη θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τόσο ώστε να χρηματοδοτηθεί αυτή η νέα παγκόσμια εταιρική σχέση βρίσκοντας μια ισχυρή ισορροπία ανάμεσα στις τρεις διαστάσεις οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον τι τρει διαστάσεις της βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, θέλουμε να προωθήσουμε συνεκτικές πολιτικές και να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τους στόχου μας και τα αποτελέσματα που θα πρέπει να επιτύχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι. Το τελικό κείμενο της διάσκεψης κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να σχετίζεται με τη μεσοπρόθεσμη εφαρμογή των στόχων για το πρόγραμμα μετά το 2015 ε, που θα εγκριθεί και στη Νέα Υόρκη το Δεκέμβρη ε, του 2015. Θα χρειαστούμε έτσι λοιπόν για το COP21 μία ισχυρή βάση ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία πλαίσιο για τις ε, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και τη σχετική διάσκεψη στο Παρίσι το Δεκέμβρη οι δημόσιοι πορεί, οι ιδιωτικοί ποροί, τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, ε, όλα αυτά τα μέσα θα πρέπει να συνδυαστούν με τα μη οικονομικά μέσα υλοποίηση των στόχων μας. Όντως είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τις επενδύσεις, να ενισχύσουμε τις θεσμικέ δυνατότητες που έχουμε, να τονώσουμε το εμπόριο και τις επενδύσεις, να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και να ενθαρρύνουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Ε, πέραν αυτού, αυτή είναι η νέα σχέση προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο παρακολούθησης, ευθύνης και αξιολόγησης ε, που θα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του προγράμματος ε, για την περίοδο μετά το 2015. το, το τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο θα πρέπει να συνδυαστούν και να συνεργαστούν οι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί εταιροί για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Κυρίες και κύριοι, είναι αποφασισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να διαδραματίσουν έναν ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο σε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ε, μεριμνώντας ώστε να υπάρξει σύγκληση των θέσεων. Η διάσκεψη 26ης Μαΐου ε, οδήγησε σε μια θέση για τη δημόσια στήριξη, ε, όπου επιβεβαιώνεται η δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών να φτάσουν το ποσοστό το 0,7% του ΑΕΠ ε, για την ε, δημόσια χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή βοήθεια για το πρόγραμμα για την περίοδο μετά το 2015 καθώς και την προτεραιότητά τους υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών θα πρέπει να διευκολύνουν επίσης ε, την εργότερη συμμετοχή της Ένωσης και των κρατών της στις προϊόντες διεθνείς διαπραγματεύσεις ώστε να τελεσφορήσουν. Η επιτυχία αυτής της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης είναι συνάρτηση της συμβολής όλων όλων μας ε, είμαι πως θα αποφασισμένοι, θα διαδραματίσουμε το ρόλο μας και θα συνεργαστούμε επικοδομητικά με όλους τους συνομιλητές μας και κυρίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τρόπο ώστε να μπορέσουμε να καταρτήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα για την περίοδο μετά το 2015, ένα πρόγραμμα φιλόδοξο που θα οδηγήσει σε μεταρρυθμίσεις αλλά και σε ολοκλήρωση των πολιτικών μας. Αυτό δηλαδή που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Υπουργέ και τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Επίτροπος Μίμητσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ. Μία εβδομάδα έχουμε μόνο μέχρι τη διάσκεψη του ΟΗΕ στην Αντισαμπέμπα για τη χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτά και για την σχετική έκθεση του Κοινοβουλίου για την φοροαπαφυγή και την φοροδιαφυγή αποτελούν τα θέματα αυτά προτεραιότητα για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι για την εξασφάλιση της επιτυχίας της διάσκεψης, γιατί θα είναι κρίσιμο και για την διάσκεψη της Νέας Υόρκης και για την διάσκεψη των Παρισίων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και με ευγνώμων για την ε, μεγάλη δέσμευση του Κοινοβουλίου στην ε, προπαρασκευαστική αυτή περίοδο σε ό,τι αφορά και την διάσκεψη για την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και για την ατζέντα μετά το 2015 και χαίρομαι που έξι από εσάς θα συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ε, συμμετάσχουν στην διάσκεψη. Ο πρόεδρος Γιούνκερ, όπω είπατε, εκπρόσωπος Μογκερίνη και εγώ θα εκπροσωπήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αντίσα μαζί με τους εκπροσώπους των εθνικών κυβερνήσεων θα εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να μιλούν με μία φωνή σε αυτές τις τελευταίες και κρίσιμες φάσεις. Θα ήθελα να σας εξηγήσω ποιες είναι οι γενικότερες αρχές και προσδοκίες σύμφωνα με τις οποίες θα κινηθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει μία μεταμόρφωση και χρειάζεται μία φιλόδοξη δέσμευση που θα καλύψει, καλύψει όλα τα επίπεδα ε, επενδύσεων σε ό,τι αφορά και τις ε, εφαρμογή. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ένα πιο στρατηγικό ρόλο για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια προκειμένου να υπάρξει μόχλευση και αξιοποίηση πλήρης του δυναμικού. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει καθολικότητα. Τελείωσαν οι μέρες διάκρισης βορράς και νότου. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική εταιρική σχέση για να πετύχουμε την ατζέντα μας και θα πρέπει κάθε χώρα να συνδράμει αυτό που της αναλογεί και ο ιδιωτικό τομέα και η κοινωνία των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να δραματίσει το ρόλο της στο εσωτερικό της και με τις εξωτερικές της δράσεις. Κατά τρίτον, το συνέδριο θα πρέπει, η συνέλευση θα πρέπει να προωθήσει ένα ε, διαφανές και αξιόπιστο πλαίσιο για να μπορέσουμε να παρακολουθούμε όχι μόνο τις οικονομικές μας δεσμεύσεις, αλλά και τη συνολική πρόοδο για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλοι έχουμε εργαστεί σκληρά για να πετύχουμε ένα φιλόδοξο έγγραφο στη διεθνή διάσκεψη που θα ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες ε, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 26 Μαΐου. Ήταν πραγματικά μεγάλη πρόκληση, μεγάλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στις διαπραγματεύσεις. Το τελευταίο κείμενο ε, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί το έγγραφο και εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες και διαφορές και σε ό,τι αφορά την διάσκεψη για το τι θα γίνει μετά το 2015. Συνεχίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι διαπραγματεύσει και ενδεχομένω να συνεχιστούν και στην Αντίσα Μπέμπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διδραματίσει το ρόλο που τη αναλογεί σε ό,τι αφορά τη φιλοδοξία των διαπραγματεύσεων και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. 58 εκατομμύρια ευρώ επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγαλύτερο δωρετή παγκοσμίω έχουμε εκ δεσμευθεί για να πετύχουμε τους στόχους του 0,7% σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ και σε ό,τι αφορά την ατζέντα από το 2015 συμπεριλαμβανομένων μιας πιο φιλοδοξής προσπάθειας για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Δυστυχώς αυτή η δέσμευση δεν έχει ακολουθηθεί από άλλους μεγάλους δωρητές. πάνω από 100 δις ευρώ θα κινητοποιήσει όπως εκτιμάται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει η ανάλογη επένδυση στις ε, χώρες που χρειάζεται. Με μόχλευση έως και 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 16 δις ευρώ θα αφιερωθούν για την αλλαγή του κλίματος και στους σχετικούς στόχους και 35 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μια, ένας υπολογισμός της ετήσιας αξίας των εξαγωγών των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τέλη και χωρίς προσωστώσεις, αγαπητοί βουλευτές. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τώρα την έκθεση του Κοινοβουλίου για την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη γενική ανάλυση της πολύ συνεπτικής αυτής έκθεσης. Έχοντα συνταλλάξει απόψει με την εισηγητή κυρία Σλάν σε διάφορε περιστάσει, αντιλαμβάνομαι τη σημασία του που αποδίδει το Κοινοβούλιο στα θέματα αυτά και σημειώνω με προσοχή τις ε, προτάσεις σας, το σχέδιο δράση σα για την υποστήριξη των αντίστοιχων χωρών για την κινητοποίηση πιο πολλών εγχώριων πόρων. Η καλύτερη κινητοποίηση των εγχώριων πόρων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά τις πιο αξιόπιστες κρατικές δαπάνες και στις πιο σωστές αξιοποίηση της διοικητικής ικανότητας των χωρών αυτών. Η χρήση των εγχώριων αυτών πόρων και η καταπολέμηση της προδιαφύγης προαποφύγης και των παράνομων ροών κεφαλαίου είναι σημαντικά στοιχεία και θα συζητηθούν στην Αντισαμπέμπα. Η διαπραγματεύσεις για το έγγραφο της Αντισαμπέμπα ήταν πολύ περιπλοκές. Και το τελευταίο έγγραφο θεωρούμε ότι αποτελεί ένα καλό συμβιβασμό που αποτυπώνει πολλά, τα πιο πολλά από τα θέματα που περιλαμβάνονται και στην έκθεση του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν ακόμα δυσκολίες για την Επιτροπή του ΟΗΕ, για την φορολογία και το σχετικό διακυβερνητικό σώμα. Υποστηρίζουμε το να δώσουμε μεγαλύτερη φωνή και ρόλο στις αναπτυσσόμενες χώρες για τον ορισμό της ατζέντα αυτής χωρίς να, να δημιουργήσουμε άλλο ένα αντικυβερνητικό σώμα απαραίτητα. Να επικεντρωθούμε στην ουσία και όχι να λαμβάνουμε αποφάσει για την μορφή στην παρούσα φάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα υποστηρίξουν αυτό το δύσκολο μονοπάτι στα πλαίσια μιας παγκόσμιας δερικής σχέσης. Θα υπάρξει και ένα σχετικό έγγραφο με τον τίτλο Collect More, Spend Better. Αγαπητοί βουλευτέ, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να πετύχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να το πάρουμε ω δεδομένο όμω. Στην Αντίσα θα έχουμε μία μοναδική ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε την παγκόσμια συνεργασία για τα επόμενα χρόνια. Ας φροντίσουμε να έχει σημασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Και τώρα για την Επιτροπή ΕΚΟΝ, ο κύριος Μπαγιέ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη δουλειά που και για το γεγονό ότι έλαβε υπόψη τι προτεραιότητε τη Επιτροπή ΕΚΟΝ. Η φοροδιαφυγή είναι μάστιγα, ε, χάνουν πόρου στα κράτη και μπορεί να επηρεάσει αυτό το σύνολο των πληθυσμών, γιατί έχει να κάνει με την κοινωνική προστασία, την απασχόληση, την υγεία, την εκπαίδευση κτλ. Γι' αυτό η Κομισιόν θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τρει προτεραιότητε. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των ε, φορολογικών διοικήσεων, ώστε να εισπράττονται δίκαιοι φόροι. Θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της φορολογικής βάσης στις χώρε χώρες ε, μέσω πρωτοβουλειών όπως το BEPS, αναθεωρούντας τη σύμβαση της διπλής φορολογίας και τρίτον θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αρχή της καλής διακυβέρνησης και της φορολογικής δικαιοσύνης. Θα πρέπει να, δείξουμε επίσης, ε, εμείς, να δώσουμε επίσης εμείς το παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να δουλεύουμε με ε, ενδιαμέσου ας πούμε σε φορολογικούς ε, παραδείσους για να δημιουργήσουμε αντί για φαύλους κύκλους ε, υγιείς κύκλους για να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Τώρα θα μιλήσουν εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Ρούμπικ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την συνάδελφο ε, Σλάιν για την καλή συνεργασία και την καλή αντιμετώπιση. Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι καταβάλουμε προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια στην αναπτυσσόμενη πολιτική, να θέσουμε, στην πολιτική ανάπτυξη να θέσουμε νέα πρότυπα. Αλλά αυτό που λένε και πολλές κυβερνήσεις ε, στον κόσμο μας ε, κάνει να σκεφτούμε πού είναι οι αιτίες, πού είναι τα αίτια. Έχουμε πρόσφυγες, έχουμε μετανάστες και δεν υπάρχει ανάλυση του τι προκαλεί τα προβλήματα αυτά, ποια είναι τα αίτια και ότι δεν υπάρχει ανάλυση της φτώχειας. Γιατί υπάρχει φτώχεια, γιατί έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Η ανεργία εξαγάγεται στην Ευρώπη. Και εμείς, εν μέρη, ξαναδίνουμε τα λεφτά αυτά τα οποία βγάζουν οι μετανάστες στις χώρες μας, στις χώρες αναπτυσσόμενες. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι με τους κανονισμούς του ΠΟΕ, το Everything But Arms, κοιτάμε τι γίνεται με τα όπλα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν και οικογενειακές επιχειρήσεις. Το βασικό είναι να μην αποστέλλετε χρήματα. Η έννοια της συνεργασίας θα πρέπει να ενισχυθεί η εκπαίδευση, η παραγωγή ενέργεια σε, σε τοπικό επίπεδο και όλα αυτά θα μα βοηθήσουν στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία να έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε και Υπουργέ, για όλα όσα είπατε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συμφωνία την επόμενη εβδομάδα στην Τσαμπέμπα και οι συζητήσει σήμερα στην Νέα Υόρκη ελπίζω να είναι γιατί θα θέσουν την ημερήσια διάταξη και για την Νέα Υόρκη και για το Παρίσι. Ε, εάν τα πάμε καλά εκεί, στις επόμενες διασκέψεις θα δυσκολευτούμε περισσότερο. Ε, ξεκαθαρίσαμε την θέση μας στην έκθεση Περέιρα για την αναπτυξιακή βοήθεια. Εγώ θα μιλήσω τώρα για το φόρο. Ο ΣΑΕΚ τιμάει ότι αν αυξήσουμε την, τα φορολογικά έσοδα κατά 1% εκατό αναπτυσσόμενες χώρες θα διπλασιάσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα τα σαν διπλασιάζαμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Άρα η φόρη είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τα φορολογικά προβλήματα. Θα πρέπει και οι εταιρείε και οι, τα άτομα να πληρώνουν όσο τους αναλογούν. Να σταματήσουμε τι παράνομε πρακτικέ όπως τα ελείποντα ας πούμε τιμολόγια των εταιριών ή οι λαθροχειρίες με τα τιμολόγια ούτως ώστε να μην πληρώνουν κάποιοι τους φόρους τους. Επίσης υπάρχουν τρομακτικά νούμερα. Ε, στην υποσαχάρια Αφρική 50 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο χάνονται ε, σε φόρους που δεν πληρώνονται. Αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να είχαν πληρώσει ε, υγειονομική περίθαλψη, ε, φροντίδα των παιδιών, ε, να μην υπάρχει κακή διατροφή και αυτοί που αποφεύγουν να πληρώνουν τους φόρους τους, στην πραγματικότητα βγάζουν το φαγητό από το στόμα των παιδιών. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις, ακούσαμε μερικές σήμερα και χρειαζόμαστε και νέους λόγους λογοδοσίας, ε, εκθέσεις αναχώρα, δημόσιες. Θα πρέπει να υπάρχουν δημόσια αρχεία για το τι κάνουν αυτές οι χώρες, ούτως ώστε να εντοπίσουμε αυτούς που δεν πληρώνουν. Αυτά θα πρέπει να συζητηθούν σε επόμενες συζητήσει. Ευχαριστώ. Κυρίω Γκέρικε. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη Επιτρόπη Μίμητσα. Είπατε ότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερο δωρητή αναπτυξιακή βοήθεια. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο με τα μέτρα μα ε, πετυχαίνουμε του στόχου που αναλογούν στι επενδύσει μα. Όχι, είναι η απάντηση. Ω συντονιστή του ECR για την αντιπροσωπεία και Ήμουν στην κοινοβουλευτική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ και μίλησα με συναδέλφους από τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Μας λένε ότι η Ευρώπη είναι δύσκολος εταίρος. Είμαστε μη ρεαλιστές στις αξιώσεις μας σε ό,τι αφορά τα θέματα και υποχρέωση για τον ε, εκπρόσωπο στα θέματα φύλου. Όταν μιλάμε για θέματα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, ε, είναι σημαντικό αυτό. Μίλησα με πολλούς ε, ε, εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας που είναι θυμωμένοι σε ό,τι αφορά τους φόρους τους ε, γιατί χάνονται τεράστια ποσά ετησίως από την ελληπή συλλογή φόρων και ζητώ ένα ειδικό πρόγραμμα για το 2020 με τον στόχο του 2020 να υπάρχουν ναι, σε οικονομικές δομές και τι διακόπτη πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Μπεθέρα, Υπουργέ, Επίτροπε, το Σεπτέμβριο του 2002 ο Μάριο Δράγκη φόβησε τους ε, επενδυτές με τη διαβόητη φράση whatever it takes, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Ε, υπήρξαν πάρα πολλές πολεμικές στη Γερμανία όπως έλεγαν, που έλεγαν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν κατά των συνθήκων. Το Ευρωπαϊκό, Κοινοβου... το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, είπε ότι επιτρέπει στην ΕΚΤ να, να αγοράσει ε, ομόλογα για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Όταν μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα ε, στα Νησάμπεπα μεθόδους χρηματοδότησης, ο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για να προσδιορίσουμε την ε, συνεργασία για την ανάπτυξη και τις πολιτικές ανάπτυξης, ε, μιλώντας για τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ε, δημιουργούν το 90% των, ε, ε, της οικονομίας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων, όταν μιλήσουμε για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όταν ε, μιλήσουμε για το πώς θα πληρώσουμε για την φιλόδοξη ατζέντα ε, τα επόμενα 15 χρόνια, να μην ξεχνάμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας που έλεγε το 2008 ότι στα πλαίσια της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη θα πρέπει να υλοποιήσουμε δράσεις εξωτερικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. δημοκρατία, κράτος δικαίου, καθολικότητα και το αδιέρετο των ε, ανθρωπίνων ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει την διαδικασία δημιουργίας ενός ε, εργαλείου δεσμευτικού διεθνούς για να προωθήσουμε ε, λύσεις για τα θύματα σε περίπτωση που οι εθνικές δικαστικές αρχές δεν μπορούν να τιμωρήσουν τους ενόχους εταιρείε πολυεθνικές κτλ. Όταν μιλάτε σας παρακαλώ πρέπει να μιλάτε πιο λογικά γιατί αλλιώς το μήνυμά σας δεν θα περάσει. Δεν μπορώ να σας διερμηνεύσω διερμηνείς με αυτή την ταχύτητα. κυρία Σάντσες Καλντέντι. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, συμφωνώ με την κυρία Μακάβαν και με άλλους συναδέλφους ότι η ίσπραξη των φόρων είναι το κλειδί για όλα αυτά. Για κάθε ευρώ που λαμβάνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες μέσω των εμβασμάτων των μεταναστών, μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων, χάνουν δύο ευρώ ε, λόγω ε, παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, ε, περίπλοκων λογιστικών, ή το γεγονός ή λόγω του ότι πληρώνουν ε, ε, λόγω του δημόσιου χρέους. Ε, εμείς όταν μιλάμε δεν μιλάμε με μια συνέπεια. Θα πρέπει να υπάρχει ε, σωστή ε, φορολογία και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Θα πρέπει επίσης να μην πληρώνονται αβίω, αβίωτα τοκοχρεωλήσια ή παράνομα ε, για το δημόσιο χρέος. Ε, σήμερα στην Ευρώπη μας δίνεται μια ευκαιρία να είμαστε συνεπείς. Ε, θα πρέπει όμως να υπάρχει γι' αυτό και η πολιτική βούληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, μία μελέτη που αναφέρεται και στην έκθεση της κυρίας Λάιν καταδεικνύει ότι οι φορολογικοί καθόντε, κανόνες στην Ολλανδία από που και προέρχομαι κοστίζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες 150-155 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την ρόλο μας ως δωρητές αναπτυσσόμενης βοήθειας, αλλά κάθε ευρώ που δεν δίνεται στην Αφρική για δουλειά που λαμβάνει η χώρα εκεί είναι ε, ένα ευρώ που αφαιρείται από την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνουμε. Ζητήσαμε λοιπόν να υπάρξει ένα δημόσιο μητρό στο οποίο θα μπορούμε να δούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης κάθε εταιρείας, ο πραγματικός ε, ιδιοκτήτης, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει φορά που φύγει και φροντιαφυγή εκ μέρους των επιχειρήσεων. Μπορούμε να μιλήσουμε όσο θέλουμε στην Αντισαμπέμπα. Αν εξακολουθήσουμε να επιτρέπουμε τα ψώνια από πλευρά των επιχειρήσεων χώρου φορολόγησης δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε στην υποσαχάρια Αφρική σε επίπεδο, στο επιθυμητό επίπεδο ούτε την εκπαίδευση, ούτε την υγεία, ούτε τίποτε άλλο. Άρα θα ζητήσω από να πολεμήσει την Αντισαμπέμπα για μια καλή νομοθεσία για την φορολογία. Ευχαριστώ. Κύριε Σκοράου, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντα συγχαρητήρια στη συνάδελφη για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε για μια έκθεση που είναι πραγματικά σημαντική. Πολύ σωστά αυτά που είπε η κυρία Μακάβαν. Όταν μιλάμε για τόσα λεφτά, για δισεκατομμύρια τα οποία εξαφανίζονται, αν είχαμε ένα καλό σύστημα καταπολέμησης φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, θα τα είχαμε αυτά τα λεφτά και θα μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε, όλη αυτή την πολιτική που θέλουμε. Πρέπει να βρούμε τα οικονομικά εργαλεία για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη. Αν υπήρχε καλό επίπεδο καταπολέμησης της φοροαποφυγής θα είχαμε όλα αυτά τα εργαλεία. Ε, οι εκθέσει αυτέ είναι πολύ σημαντικές. Είναι ένα καλό κίνητρο. Ε, αυτό το σύστημα country by country, ε, τεχνική βοήθεια στις χώρες, ε, ακόμη και η δημιουργία μιας διακυβερνητικής οργάνωσης. Και αυτό που είπε η συγγήτρια. Ελπίζω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, θα γίνει, θα περάσει και μετά θα περάσει και από την Ολομέλεια, έτσι με ε, μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ ο Στυρ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Με την επόμενη διάσκεψη του ΟΗΕ για τη χρηματοδότηση ε, στην Αντίσα και την σύνοδο στη, Νέα Υόρκη καθώς και την COP21 στο Παρίσι θα πρέπει να επαναλάβουμε το μήνυμα που στείλαμε τον Απρίλιο όταν εγκρίναμε το ψήφισμα του κυρίου Περέιρα βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει το ρόλο της ως βασικός δωρητής Όμως ε, θα πρέπει κάποιες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο της ευθύνης διότι δεν υπάρχει κανένας άλλος που να αφιερώνει 0,7% του ΑΕΠ για την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να αρχίσουμε να επενδύουμε σε παραγωγικούς τομείς που θα είναι κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη, για την ε, τον εγχώριο και τον ε, ε, τομέα για τις εγχώριες και για τις ξένες επενδύσεις. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερες φορολογικές αρχές. Αυτό είναι βασικό στοιχείο στην πολιτική μας ε, και γι' αυτό θα υποστηρίξω την έκθεση του κυρίου Σλάιν για την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να επικεντρωθεί ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων για την φοροσυλλογή αλλά και για την εκρίζωση της ακραίας φτώχειας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε νέα προγράμματα και θα πρέπει να στεφθεί με επιτυχία η διάσκεψη Αντίσα Κύριο Σίλβα Περέιρα, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή διακυβεύεται στη διάσκεψη της Αντίσα Μπέμπα για την ε, χρηματοδότηση της ανάπτυξης ε, που αρχίζει σε λίγες ημέρες. Ε, διακυβεύεται κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι η κινητοποίηση των επαρκών κονδυλίων ώστε να εφαρμόσουμε την το παγκόσμιο με ε, αναπτυξιακό θεματολόγιο από το 2015 έως το 2030. Είναι απαραίτητο η διεθνής κοινότητα να καταλήξει σε μια φιλόδοξη συμφωνία στην Αντίσα Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη με σαφήνεια προσδιορίσε τη θέση του και συμπεριέλαβε ε, το στόχο 0,7% του ΑΕΠ ε, για να διοχετευτεί στην αναπτυξιακή βοήθεια και επίσης ε, αναφέρθηκε σε ένα χρονοδιάγραμμα και ξέρουμε όλοι ε, πως δυστυχώς η θέση του Συμβουλίου δεν στάθη στο ύψος των περιστάσεων. Με τις προπαρασκευαστικές εργασίες της διάσκεψης της Αντίσα βλέπουμε και άλλα ανησυχητικά στοιχεία. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ακόμη μικρότερη διαθεσιμότητα των υπολείπων εταίρων για συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις. Θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες και στις αναδυόμενες οικονομίες για να υπομισθούν τη δική τους ευθύνη. Διότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις από πλευρά τους. Η διάσκεψη της Αντίσα θα πρέπει να είναι η διάσκεψη της ευθύνη σε σχέση με την δημόσια χρηματοδότηση αλλά και για το αναπτυξιακό θεματολογικό. Γι' αυτό υποστηρίζουμε ε, ε, την ε, έκθεση του κυρίου Σλάιν για την ε, διεθνή συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Σας ευχαριστούμε κυρία Χαουταλά. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Όλο ένα και περισσότερες ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μας λένε ότι θέλουν να διαρρήξουν αυτό το δεσμό εξάρτησης ε, από την αναπτυξιακή βοήθεια. Στη Ζάμπια παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια ανέρχεται μόνο στο 2,5% του ΑΕΠ. Ε, όμως Υπάρχει και μια συγκεκριμένη ανάγκη για αυτές τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες να μπορέσουν δηλαδή να συγκεντρώσουν, να ομοδοποιήσουν την αναπτυξιακή βοήθεια. Μπορούμε να βελτιώσουμε επίσης ε, την ε, συλλογή φόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γι' αυτό όμως χρειάζεται μια σταθερική και σωστά σχεδιασμένη προσέγγιση με την Προεδρία του Λουξεμβούργου πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα λαμπρό παράδειγμα για όλες τις υπόλοιπες χώρες ως προς την ε, αναπτυξιακή χρηματοδότηση και πιστεύω ότι θα βοηθήσετε τις άλλες χώρες να υπομισθούν τις ευθύνες τους. Ε, στις σκανδιναβικές χώρες ε, πνέει ένας ψυχρός άνεμος διότι υπάρχουν περικοπές που φτάνουν μέχρι και το 40%. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, ε, Γκίλ Νέιθεν. Σας ευχαριστώ. Φαίνεται ότι ξεκινάει αυτή η έκθεση από μια λανθασμένη αρχή γιατί προσπαθούμε να απειλήσουμε περιφερειακά ζητήματα στις ε, χώρες αυτές. Αυτό της διαφθοράς είναι το βασικό ζήτημα και η Νιγηρία αποτελεί ένα κατεξήχην παράδειγμα. Αυτό δικαιολογεί και εξηγεί τη χαμηλή εμπιστοσύνη των ε, επενδυτών. Επενδύσεις σε μια χώρα με τους πιο ε, χαλαρούς ευρωλογικούς νόμους και το πιο χαλαρό ήθος. Αυτή η έλλειψη της διαφάνειας ε, είναι το κλειδί και θα πρέπει να πάψει για να υπάρχει ευθύνη. Αλλά είναι ρεαλιστικό αυτό. Έχουμε στην σημερινή εποχή τεχνολογικές εξελίξεις και αυτό είναι μια ευλογία και θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει αυτή η αξίωση, η οποία όμως είναι αντιπαραγωγική. Πρωτού αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικό τρόπο το θέμα της φοροδιαφυγής. Θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα της διαφθοράς. Αν θέλουμε να κάνουμε νομοθεσία για κάτι, ας είναι η ρίζα του κακού και όχι το παράπλευρο σύμπτωμα του κακού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βέντα, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 2015 είναι η χρονιά χρηματοδότησης των αναπτυξιακών πολιτικών. Τον Ιούλιο έχουμε τη διάσκεψη της Αντίσα Μπέμπα, το Σεπτέμβριο τα μέλη του ΟΗΕ θα συναντηθούν για να εντοπίσουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που θα αντικαταστήσουν τους στόχους της χιλιετίας μετά το 2015. Παρατηρούμε τις τάσεις αυξανόμενων αγκών των αναπτυσσομένων χωρών και τη μείωση της αναπτυξιακής βοήθειας λόγω της οικονομικής κατάστασης στις χώρες που είναι δωρήτριες. Ακούσαμε πολλά για τα οικονομικά προβλήματα και για τα φορολογικά προβλήματα, αλλά και για καινοτόμους πόρους. Οι καινοτόμοι πόροι μπορούν να βοηθήσουν να υλοποιηθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι μετά το 2015. Υπάρχει μια διεθνής οργάνωση UNIAID που με την υποστήριξη του ΟΗΕ μας πείθει πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το μοντέλο. Τα τελευταία νέα χρόνια η UNIAID μπόρεσε να χρηματοδοτήσει το 80% των αναγκών ε, των φορέων του AIDS που ήταν ανήλικοι, ε, ατόμων που είχαν επίσης ελονοσία και θυματίωση. Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσουν καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης της ανάπτυξης αυτής. Η φορολογία καθώς και η αντιμετώπιση των παράνομων οικονομικών ροών μπορεί να, βελτιω... μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των χωρών αυτών. Ο επόμενος ομιλητής ε, Νόισερ για 1,5 λεπτό. Αξιότιμη Πρόεδρε, αγάπητε Επίτροπε Μίμητσα και κυρίως ε, αξιότιμη Προεδρία του Συμβουλίου. Η Σουηδία, η Δανία, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο τι έχουν κοινό. Τι μοναδικές τέσσερις χώρες των 28 χωρών, οι οποίες έως τώρα έχουν τηρήσει την υπόσχεση για το 0,7%. Και χαίρομαι που η Προεδρία ε, του Συμβουλίου δραστηριοποιείται ενεργά εδώ στην Ολομέλεια, γιατί δεν το κάνουν αυτό όλες οι προεδρίες. Δεν έχουν επιδείξει όλες οι προεδρίες αυτή την, ε, αυτό το ενδιαφέρον για την αναπτυξιακή πολιτική. Νομίζω ότι ένα βασικό κλειδί για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας της αναπτυξιακής βρίσκεται στα αρχικά για τον κρατών μελών. Είμαι από μια χώρα, από τη Γερμανία, που είναι η πιο φτωχή, αλλά σε ό,τι αφορά το ανώτατο όριο, δεν είναι η πιο φτωχή, αλλά έχει αυξηθεί 0,4% τα τελευταία χρόνια αυτή η βοήθεια. Νομίζω ότι η Προεδρία του Λουξεμβούργου στο έτος για την ανάπτυξη θα πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να υποδείξει με το καλό της παράδειγμα ποια θα πρέπει να είναι η διεθνή συνεργασία προκειμένου να υπάρχει πιο πορεία αξιοπιστία σε διαπραγματεύσεις όπως ε, στο Παρίσι θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και δεν είναι δυνατόν σε 15 χρόνια να μην έχουμε πετύχει το ποσοστό που χρειάζεται. Ευχαριστώ κύριο Τσέλερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, σε, δύο, σε λίγες ημέρες ε, θα έχουμε ένα από τα ορόσημα στην Αντιζαμπέμπα για τους στόχους της ε, αναπτυξιακής βοήθειας για τη χρηματοδότηση των στόχων αυτών πέρα από τα οικονομικά μέτρα θα πρέπει οι χώρες οι αναπτυσσόμενες να αξιοποιήσουν τις δικές τους, τους δικούς τους πόρους για να θέσουν ένα τέλος στην πείνα και να εξασφαλίσουν μια καλή ζωή στους πολίτες τους. Τα αναπτυσσόμενα κράτη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να αυξήσουν την συλλογή φόρων. Γιατί είναι πλούσια θα τα κράτη σε πόρους, σε νέους, σε ένα οικονομικό δυναμικό για βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά δεν μπορούν τα χρήματα αυτά να καταλήγουν στις τσέπες των λίγων και να βγάζουν τα κέρδη εκτός χώρας ε, οι διεθνείς ε, εταιρείες. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα δημόσιο σύστημα και ένα τέτοιο για να επιλύονται τα προβλήματα επιτόπου. Και θα πρέπει η διεθνή συνεργασία σε θέματα φορολογικά να προωθηθεί. Και η έκθεσή μας ε, δίνει βασικά κίνητρα προς την κατεύθυνση, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν και στην πράξη. Ευχαριστώ. Yes, thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λίτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε στα G77 μία εβδομάδα πριν ε, την Αντισαβέμπα δεν υπάρχει συμφωνία. Και έτσι μειώνονται οι πιθανότητες επιτυχίας της Αντισαβέμπα. Γι' αυτό σε ζητούμε ως σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σκεφτούν όλοι τη στάση τους στη διάσκεψη. Και αυτό αφορά και το 0,7% ως δέσμευση από τις ε, βιομηχανικές χώρες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτό το 2030 για να εκπληρώσουμε αυτή την δέσμευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρηματοδότηση παίζει σημαντικό ρόλο. Για την μελλοντική διάσκεψη στην Αντίσα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου τα αποτέλεσμα να αποτελέσουν ορόσημο στην αναπτυξιακή πολιτική. Και θα ήθελα όλοι όσοι συμμετέχουν. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους θα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στη διαδικασία του Catch the Eye. πρόεδρος, πρώτος ομιλητής, ο κ. Μισελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα μεγάλη προσοχή τη συζήτηση και έχω μια συγκεκριμένη πρόταση να κάνω. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να προτείνουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι συγκεκριμένα προγράμματα για το πώς θα συλλέγουν φόρους. Πέρα από την χρηματοδοτική βοήθεια και την παράσχεση τεχνογνωσίας, ε, αν τους δώσουμε εμπειρογνώμονες για το, που θα τους βοηθήσουν να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή, ε, θα είναι πολύ καλό. Μπορούμε να προσφέρουμε τέτοια προγράμματα στις ε, χώρες και επίση, ε, μην ξεχνάτε ότι δίνουμε και τέτοια προγράμματα στι χώρε που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όχι λοιπόν και στι αναπτυσσόμενε χώρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να προτείνουμε πιο συγκεκριμένα μέτρα σε αυτέ τι χώρε και να τι βοηθήσουμε να καταπολεμήσουν την φοροδιαφυγή. Ένα ακόμα σχόλιο. Η φοροδιαφυγή δεν σημαίνει να μην υπάρχουν να υπάρχουν μάλλον ψηλοί φόροι. Ε, αντίθετα, θα πρέπει να, έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν και χαμηλού φόρου αν χρειάζονται αυτέ οι χώρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει η κυρία Ζαμπόφσκα. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε ζήσει το θέμα της υπερβολικής χρέωση, όχι μόνο ως θέμα των αναπτυσσόμενων χωρών. Ο συνδυασμός του λαϊκισμού και της υπερβολικής ε, χρέωσης έφερε ε, σε δύσκολη κατάσταση και ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. υπερβολικά χρέη που γονατίζουν την οικονομία και δεν ε, μένει ενέργεια για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Και αυτή τη χρέωση οδηγεί σε μόνο σε εκ νέου χρέωση. Η μοναδική ε, δυνατότητα είναι οι συζητήσει μεταξύ των πιστωτών και των ε, ε, χωρών. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει και για την Αιθιοπία αλλά και για την Ελλάδα. Η βασική προϋπόθεση είναι όμως ότι θα πρέπει οι όσοι χρωστούν να προφέρουν τις ευθύνες τους και να μην διοργανώνουν δημοψηφίσματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Κυρία Πρόεδρε, η τεράστια φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη διακυβέρνηση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο μέσος λόγος των φόρων προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ιδιαίτερα χαμηλός και κινείται μεταξύ 10% και 20%. Έτσι, οι αναπτυσσόμενες χώρες αδυνατούν να φορολογήσουν τα κέρδη των πολυεθνικών που αναπτύσσουν κερδοφόρες δραστηριότητες στο έδαφος τους αυτό σημαίνει απώλεια τεράστιων φορολογικών εσόδων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων του κράτους. για το λόγο αυτό οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται εκεί όπου πραγματοποιούνται τα κέρδη. όμως οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν πρόκειται να μπουν στον δρόμο της ανάπτυξης όσο βαρύνονται με το άχθος του τεράστιου δημοσίου χρέους τους. για το λόγο αυτό πρέπει να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή το ψήφισμα του οηε του σεπτεμβρίου του 2014 για τη διαγραφή του κρατικού χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μας μιλούσε ο Επίτροπος για μια συνεκτική γραμμή ως προς το ε, οικονομικό περιβάλλον ε, για την, την αρχή της οικουμενικότητας ε, ως προς την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε για το ποσοστό του 0,7% του ΑΕΠ. Δεν έχει αναλυθεί τέτοια δέσμευση από όλα τα μέρη και ενδιαφέρονται όλα αυτά που μας είπατε, όμως δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε τη σημασία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι συχνά τίθεται αυτό το ζήτημα σε αυτές τις χώρες και οι χώρες τις οποίες στέλνουμε αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια συχνά παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να συνδέσουμε την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας με την τήρηση οικουμενικών αρχών και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ, Επίτροπε, για τα φιλόδοξα σχέδια που έχετε για την διάσκεψη στην Αντίσα Μπέμπα. Προωθείτε ένα συνεκτικό πρόγραμμα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ηγετικό ρόλο για την παροχή ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Μην ξεχνάμε όμως ότι δεν είναι μέσω αυτό για την εκρίζωση της ευτόχειας. Γι' αυτό θα χρειαζόμασταν μια πιο κοινοτόμα πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και να υπάρχει κατάλληλη συνεργασία με τους εταίρους μας ούτως ώστε να ευοδοθούν οι προσπάθειές μας. Όπως λέει και ο κύριος Λάιν, ε, είναι απαραίτητο να καταπολεμήσουμε τη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους για να μπορέσουν και αυτές οι ίδιες οι χώρες να αναπτυχθούν. Σας ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος Μίμητσα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δίνετε, δείχνετε για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής ατζέντα, για την διάσκεψη της Αντισαμπέμπα, για τις ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις σας. Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει ψηλή φιλοδοξία και να δεσμευτεί να συνεχίσει την αναπτυξιακή βοήθεια και να εφαρμόσει τους στόχους για την ανάπτυξη. Επίσης σχολιάσατε θέματα πέραν τη αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια αυτά. Εκεί μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο μετά το 2015. Για το θέμα της παρακολούθησης και του follow-up θα πρέπει να παραμείνουμε φιλόδοξοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ένα, μια προσπάθεια ετήσια φιλόδοξη ε, λογοδοσίας για να παρακολουθήσει την πρόοδο. Το 2015 δημοσιεύσαμε τις εκθέσεις τον περασμένο μήνα. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς μπορούμε να ισχύσουμε αυτή τη διαδικασία στα πλαίσια μιας παρακολούθησης και λογοδοσίας μετά το 2015. Ήδη σε αυτή τη φάση θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει την εφαρμογή της χρηματοδότησης της ανάπτυξης μετά το 2015 και πώς θα εφαρμόσει το θεματολόγιο για την ανάπτυξη. Εξετάζουμε προσεκτικά πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές της ε, θα πρέπει ίσως να τις αναθεωρήσει για να προωθήσει πλέον το νέο θεματολόγιο. Η αρχή της ε, συνεπούς πολιτικής για την ανάπτυξη είναι πολύ πιο σημαντική τώρα παρά ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να προωθήσει διάφορες δράσεις για να προωθήσει το θεματολόγιο το 2015. Αυτό σημαίνει πλήρη ε, προσέγγιση, υποστήριξη των, υποστήριξη των αναπτυσσομένων χωρών για να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Θα προωθήσουμε τις δράσεις που προωθεί το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του ε, θα τις, αφού τις σκεφτούμε και μας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί σας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε. Ο Υπουργός Σμιτ έχει τώρα το λόγο. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την τον εισηγητή, συγγνώμη, διότι χάρη σε αυτή την έκθεση μπορέσαμε να έχουμε ένα καλό εφαλτηρίο για τη συζήτηση που πρέπει να γίνει προπαρασκευαστικά πριν από την σύνοδο στην Αντίσα Μπέμπα. Όπως τόνισε και ο Επίτροπος, έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει σε παγκόσμια κλίμακα η προσπάθεια. Με τις παρεμβάσεις που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, διαπιστώνουμε και επιβεβαιώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν ξεκάθαρη θέση ως προς το στόχο της διάσκεψης. Ο στόχος δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην παροχή της αναπτυξιακής βοήθειας. Οφείλουμε να επιμείνουμε σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, χρησιμοποίηση δε όλων των διαθέσιμων πόρων οικονομικών και άλλων. Η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να παραμείνει βασική πηγή χρηματοδότησης, κυρίως για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και για τις ευάλωτες χώρες, υπό την αίρεση και το τονίζω ότι θα είναι καλά εστιασμένη και ε, ότι θα υπάρξει και μια χρηστή ε, διαχείριση αυτής της αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε και σίγουρα η εκπαίδευση είναι βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής πολιτικής, το ίδιο και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. ή επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας ε, είναι ένα άλλο ε, απαραίτητο κομμάτι της αναπτυξιακής βοήθειας ε, και μην ξεχνάμε και ε, τη, τα μικροδάνεια και άλλους αναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων σε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι αμέριστη η δέσμευση που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη για να τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας ε, και για να είναι πραγματικά πρόσφορη η πολιτική μας και να οδηγήσει στη δημιουργία μιας ουσιαστικής παγκόσμιας εταιρικής σχέσης. Σας ευχαριστούμε και τώρα η κυρία Σλάιν. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ε, καλή του διάθεση. Αυτός τους μήνες μας ε, έδειξε ότι μπορεί να συζητήσει, έλαβε υπόψη του επίσης τις προτάσεις μας. Πολύ καλό αυτό. Πολλές φορές συζητήσαμε και ξέρει ότι είμαστε πεπισμένοι ότι η δημιουργία ενός ε, διακυβερνητικού οργανισμού ε, είναι ο μόνος τρόπος να υπάρχει σωστή εκπροσώπηση και των αναπτυσσομένων χωρών. Έχουμε τη UN Taxation ε, Committee. Σήμερα αυτή έχει 25 μέλη. Είναι σημαντικό ποιος συμμετέχει εκεί και ποιος μιλάει εν ονόμα της κυβέρνησής τους. Μερικές φορές επίσης ο τύπος είναι ουσία. Ελπίζω λοιπόν η αυριανή ε, ψήφος θα μας βοηθήσει για να απομπλέξουμε την ε, συζήτηση για να φτάσουμε σε αυτό φιλόδοξο κείμενο στην Αντισαμπέπα. Ευχαριστώ το Συμβούλιο, ευχαριστώ την Πρόεδρο Μακάβαν που θύμισε ότι το Country by Country Report η αναχώρα ε, εκθέσεις είναι σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Είναι βασικό στοιχείο του σχεδίου δράσης και ελπίζω ε, αύριο όλες οι ομάδες να μας υποστηρίξουν για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που εισέφεραν στη συζήτηση και θέλω να υπενθυμίσω ότι προφανώς υπάρχουν και πολλά πράγματα που δεν είπαμε προφορικά, αλλά υπάρχουν στο κείμενο. Δεν θέλουμε απλώς να βελτιώσουμε την κινητοποίηση των ε, εσωτερικών πόρων. Πρέπει να ε, προωθήσουμε την λογοδοσία, την ε, διαφάνεια, την διακυβέρνηση και βεβαίως πρέπει να καταπολεμήσουμε και την διαφθορά. Το λέει πολλές φορές το κείμενο. Θα πρέπει επίσης μακροπρόθεσμα να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία των χωρών αυτών, να απεξαρτηθούν επιτέλους από την εξωτερική βοήθεια. Σας ευχαριστώ και ελπίζω αύριο να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία όταν ψηφίσουμε. Thank uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Θα ψηφίσουμε αύριο. Και έχω και μια ανακοίνωση να κάνω. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ρίμουν Σερνατζότο, ο οποίο φεύγει από την ομάδα του ΕΛΚ και θα μεταβεί στην ε, ομάδα του ECR από σήμερα, 7 Ιουλίου.